Uh, Γεια σας. Αρχίζουμε. Ε, είναι πολύ βαριά η μερίσια διάταξη. Και πρέπει να σας ενημερώσουμε και για τις αποφάσεις που έλαβε η συνεδρία των συντονιστών. Θα μιλήσω πολωνικά καλύτερα. Έλεγα λοιπόν ότι ε, συνεδρίασαν οι συντονιστές και έλαβαν κάποιες αποφάσεις. Θα περιμένω λίγο να βάλετε ακουστικά, θέλετε όσοι δεν καταλαβαίνετε πολωνικά. zdecydowało w e, części e, e, Πήραμε λοιπόν αποφάσεις για διορισμούς. και για εκθέσεις πρωτοβουλίας. Μία έκθεση πρωτοβουλίας συγκεκριμένα για το ρόλο ε, ε, των θεσμικών οργανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συζήτηση αυτή η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΡΕΓΚΙ ζήτησε να συμμετέχει Αυτό το θέμα βέβαια παραμένει σε εκκρεμότητα. Άλλο θέμα, η εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εδώ οι συντονιστές ε, απέρριψαν το αίτημα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ελευθερίων. που ήθελε να είναι συναρμόδια επί της ουσίας. Διαφωνήσαμε εμείς. Συζητήσαμε και άλλα θέματα όμως στους συντονιστές, ιδιαίτερα το αίτημα ορισμένων πολιτικών ομάδων να δούμε κατά πόσο είναι θεμητές οι πρακτικές ορισμένων πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη και συγκεκριμένα ο τρόπος με τον οποίο ευθυγραμμίζονται ε, με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. E, Όλες οι πολιτικές ομάδες καλούνται να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Η κυρία Μπρέσο και ο κύριος Σόφλιν θα ηγηθούν αυτής της προσπάθειας. Οπότε, Ο ρόλος τους είναι να προετοιμάσουν ε, αυτή τη διαδικασία. Επίσης πρέπει να σας πω ότι στις 23 του μηνός έχουμε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα υποδεχθούμε τον κύριο Τίμερμανς. Στις 23 του μηνός, στις 3 το απόγευμα. Είστε όλοι φυσικά προσκεκλημένοι να συμμετέχετε στη συνεδρία σε αυτή. Ορισμένοι από εσάς ζητήσατε να καλέσουμε τον κύριο Τίμερ μας στην Επιτροπή μας. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να απαντηθούν αρχής γενομένης από την ερώτηση του κ. Σέφλιν σχετικά με τη θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτά ως προς τις ανακοινώσεις της συνεδρίας των συντονιστών. Πάμε λοιπόν στο σημείο 8 τώρα της ημερήσιας διαταξής ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, wymiany opinii. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι κάναμε μια πρώτη ταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό στις 20 του μηνός Απριλίου. Ο κύριος Ραμόν Χάουρεγγι Ατόντο είναι ο εισηγητής μας και μας ε, παρουσίασε το σχέδιο έκθεσης. Ήταν πάρα πολύ γόνιμη η συζήτηση και επικοδομητική και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Στο στάδιο του εγγράφου εργασίας βρισκόμαστε τώρα. Για το χρονοδιάγραμμα λοιπόν που προτείνεται 29 Σεπτεμβρίου αναμένουμε να συζητηθεί το σχέδιο έκθεσης που πρέπει να έχει πάει στη μετάφραση μέχρι τις 14 του μηνός. Και η τελική προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών είναι 13 Οκτωβρίου. Η εξέταση των τροπολογιών 8 listopada 2016 roku wreszcie ε, samo 5 ε, grudnia 2016. Λοιπόν, και θα ψηφίσουμε στις 5 Δεκεμβρίου. 8-11 θα συζητήσουμε τις ε, τροπολογίες. Ε, e, e, e, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ραμόν Χάουρεγγι. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο κύριος Ραμόν Χαουρεγγί, εισηγητής. Όπως μόλις μας ενημερώσατε, το έγγραφο που έχουμε στα χέρια μας για τη συζήτηση αυτή τη σημερινή είναι ένα δεύτερο έγγραφο εργασίας, τελείως άτυπο, αποκλειστικά, δεν είναι σχέδιο έκθεσης, είναι ε, ευσύνοπτο, ε, γιατί ε, υπόκειται σε περιορισμούς για τον αριθμό λέξεων. Τα έγγραφα εργασίας έχουν προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν και πρέπει να είναι πάρα πολύ σύντομα. Είναι το πρώτο λοιπόν πρόχειρο κείμενο. Θα σας πω κάποιες διορθώσεις που θα κάνω που μας στείλατε εσείς στη συζήτηση που κάναμε την πρώτη για αυτό το θέμα. Πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος ότι θα κάνουμε ένα προσχέδιο το Σεπτέμβριο και τις τροπολογίες τον Οκτώβριο και από εκεί και πέρα έχουμε προγραμματίσει την πορεία της έκθεσης για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε με το καλό το Δεκέμβριο. Πρώτον, έχω συμπεριλάβει τις δικές σας προτάσεις και από την εισαγωγή του εγγράφου έχω αφαιρέσει την πολιτική θεώρηση που ανέλυε γιατί υπάρχει πολιτική κρίση, γιατί μας έχει γυρίσει την πλάτη ο κόσμος, γιατί έχει απαξιωθεί η πολιτική, γιατί απομακρύνονται οι πολίτες, γιατί υπάρχει οικονομική κρίση. Όλα αυτά, η ε, ιδεολογική βάση της κρίσης. Ο κύριος Πρέντα πρότεινε να τα σβήσω και τα σβήσα. Γιατί προφανώς δεν ήταν αυτό το βασικό θέμα της έκθεσης. Βέβαια αυτό είναι θέμα ερμηνείας, έτσι, ο καθένας το βλέπει από τη σκοπιά του. Λοιπόν, αυτό που έκανα ήταν ότι έβγαλα όλα αυτά τα στοιχεία, τα επεξηγηματικά για τα αίτια της πολιτικής κρίσης που γνωρίζουμε. Και εκινώντας λοιπόν από αυτή την απομάκρυση του κόσμου, που σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί κανείς, αλλά φαίνεται δεν ήταν το παρόντος ή μπορεί να χωράει διάφορες ερμηνείες και πολιτικές θεωρήσεις. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που έχω να σας κάνω ε, για το έγγραφο, ότι τα έβγαλα αυτά από την εισαγωγή. Δεύτερο, μετά από αυτά που μου ζήτησε η Μπάρμπαρα Σπινέλη, Έχω συμπεριλάβει κάποια παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, ιδιαίτερα την αναφορά στην ε, Ιταλική διακήρυξη των δικαιωμάτων ε, στο διαδίκτυο του Ιουλίου του 2015, που είναι απαραίτητη αναφορά σε αυτή την εξίσωση. Ε, από τη μια έχουμε τη δημοκρατία και από την άλλη τις τεχνολογίες της επικοινωνίας, ICT. Μετά, κάτι που ζήτησε ο κύριος Άντερσον ε, των Πρασίνων, αφαίρεσα κάποιες αναφορές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρεμηνίες. Ορισμένες ε, ομάδες εκπροσώπησης τομεακής ή συντεχνιακής, τα λεγόμενα λόμπι, ομάδες συμφερόντων, μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Εγώ αυτό το είχα γράψει με κάθε καλή πρόθεση, ότι είναι πληροφορίε στη διάθεση των πολιτών. Τώρα, εάν ε, καταχρώνται ορισμένες ομάδες, ορισμένα στοιχεία και πληροφορίες και επειδή το ζήτησε ο κύριος Άντερσον, το έβγαλα και αυτό από την έκθεση. Πολλοί συνάδελφοι επίσης μίλησαν την πρώτη φορά που το συζητήσαμε και ζήτησαν να συμπεριληφθούν διάφορες ε, προτάσεις, όπως και έκανα, για μελλοντικές δράσεις και γραμμή. Ο κύριος Πρέντα επίσης ρώτησε κάτι, ε, έθεσε κάτι υπόψη μας. Η έκθεση τι φιλοδοξεί. Όχι απλώς να είναι χρήσιμη για ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και για τα εθνικά κοινοβούλια. Εμείς δεν καταθέτουμε αυτή την έκθεση στο εργασιακό μας θεσμικό περιβάλλον. Είναι ένα ανοιχτό θέμα και δεν περιορίζουμε τους αποδέκτες ποιος με ποιο τρόπο και τι θα εφαρμόσει από αυτά που εμείς προτείνουμε. Δηλαδή πολύ κάλλιστα να συνάδουν οι συστάσεις σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Έτσι απαντώ σε κάποιες αμφιβολίες που άφησε ο κύριος Πρέντα να εννοηθούν η κυρία Τέρι Κάμπρας, η κυρία Σπινέλη και η κυρία Αντινόλφη μου ζήτησαν και το έκανα να διευκολύνουμε την πρόσβαση την εκπαιδευτική και την τεχνολογική έτσι ώστε όλο και περισσότεροι να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αυτά. Αυτά γίνουν από το σχολείο για να ξεπεραστεί το χάσμα, το ψηφιακό. Υπάρχει και ο ψηφιακός αναλφαβητισμός δεν θέλουμε να ισχύει κάτι τέτοιο, να έχουμε μια μάζα ψηφιακών αναλφαβήτων ε, στην κοινωνία. Άρα δεν θέλουμε να υπάρχουν χάσματα τέτοια που να χωρίζουν τον πληθυσμό σε εκείνους που έχουν ψηφιακές δεξιότητες και σε εκείνους που τις στερούνται. Άρα θα πρέπει η τεχνολογία και η παιδεία να συνεργαστούν. Κάτι άλλο που ζήτησε η Μάιτε Παγάσα Ορθοντούα, η Μπάρμπαρα Σπινέλη, η Σαμπέλα Ντινόλφη ήταν αναφορές στην ε, εξάλληψη του ηλεκτρονικού αποκλεισμού. Δηλαδή αυτό λέγεται e-inclusion, ε, συμπερίληψη όλων στον ηλεκτρονικό κόσμο, στις τεχνολογίες πληροφορίας γιατί αν δεν επεκταθεί αυτό, αν δεν διευρυνθεί και αν δεν είναι καθολική η πρόσβαση ε, στα μέσα αυτά, πολύ δύσκολα μπορεί κάποιο να τα χρησιμοποιήσει για να έχει καλύτερη επαφή με τους κυβερνώντες. Επίσης έχω συμπεριλάβει μια αναφορά στη μεγαλύτερη ασφάλεια του διαδικτύου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία της. Η Mercedes Presso επίσης ζήτησε κάτι που πρόσθεσα, η ψηφιακή τεχνολογία να χρησιμοποιείται περισσότερο και καλύτερα στη δημόσια διαβούλευση και στις μελέτες αντικτύπου και τα λοιπά ως βοήθεια για να βελτιώνεται η διακυβέρνηση. Ο κύριος Σόφλιν επίσης και η κυρία Σπινέλη αλλά και η Σαμπέλα Ντινόλφη πρότειναν και το κάναμε να συμπεριληφθούν μηχανισμοί συμμετοχής και διάδρασης των πολιτών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που θα πρέπει να προωθούνται και όλες, όχι απλώς να ενσωματωθούν. Οι τεχνολογίες επικοινωνίας θα πρέπει να επιτρέπουν την πληροφόρηση, τη διαφάνεια, ε, την ε, συζήτηση το να εισακούεται η φωνή των πολιτών έτσι ώστε να καλυφθεί αυτό το χάσμα που υπάρχει ε, ανάμεσα στην κοινωνία και σε εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις. Να βελτιώνεται η λογοδοσία. Επίσης ο κύριος Σόπφλιν ζήτησε στο τέλος να συμπεριληφθεί η αναφορά ότι όλα αυτά να τα βλέπουμε με κάποια συγκράτηση έτσι, και να κάνουμε βήματα μικρά. Η δημοκρατία η ίδια είναι μια δυναμική ε, διεργασία και οι τεχνολογίε τη επικοινωνία θα πρέπει ε, στην αρχή να είναι αντικείμενο παρατήρηση και μετά να λαμβάνουμε μέτρα προσεκτικά να προχωράμε σιγά σιγά και όχι με βεβαιασμένε κινήσεις. Να αναρωτηθούμε κιόλας δηλαδή τι ανάγκες υπάρχουν κάθε φορά και πώς προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτά. Είμαι στη διάθεσή σας για προτάσεις. Ακόμα έγγραφο εργασίας είναι, δεν είναι ακόμα έκθεση. Το πρώτο σχέδιο έκθεσης θα το διαμορφώσουμε μαζί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, με βάση και τις δικές σας προτάσεις. ευχαριστώ. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο στους κοιόδους. Κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχήν ε, τον εισηγητή για την αναθεωρημένη πρότασή του για το έγγραφο εργασίας που μας υποβάλλει σήμερα. Είπε πολύ συγκεκριμένα ότι αυτό το νέο έγγραφο λαμβάνει υπόψη του και έχει ενσωματώσει πολλές από τις ε, παρατηρήσεις που είχαμε υποβάλει οι συνάδελφοι και εγώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ότι αναφέρει κάποιες ε, πολύ εύκολα ερμηνεύσιμες αναφορές. Αυτές δεν υπάρχουν στον δεύτερο έγγραφο εργασίας και αυτό είναι πολύ θετικό. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποια πιο σημαντικά σημεία τα οποία αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και σχεδιάζουμε την πολιτική. Σήμερα με το διαδίκτυο, με το Twitter, το Facebook και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργούν, θα πρέπει να προσαρμοστούν και τα δημοκρατικά μας πολιτεύματα νέοι τρόποι έκφρασης, νέοι τρόποι κινητοποίησης. και μία συμμετοχή στα πολιτικά με την πιο κλασική έννοια της λέξης αυτής. Θα συμφωνήσω εδώ με αυτό που είπε ο εισηγητής μιλάει για μια ψηφιακή εξέλιξη και βεβαίως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσέξουμε το θέμα αυτό και να το αναλύσουμε με κάθε προσοχή. Στο τέλος, ο εισηγητής στη σελίδα 5 αναφέρει κάποια θέματα, όπως παραδείγματο χάρη το θέμα της ορίμανσης της ψηφιακής δημοκρατίας, αυτή η μόνιμη και ενεξελίξη ηλεκτρονική δημοκρατία απαιτεί και μία συνεχή προσαρμογή του δημοκρατικού μας ε, πολιτεύματος, της ε, κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, η οποία λειτουργεί εδώ και δεκαετίες. Με μεγάλη χαρά είδα επίσης ότι η παράγραφος που αναφέρεται στα δημόσια συμφέροντα και στα ιδιωτικά συμφέροντα, σελίδα 4, έχει αναδιατυπωθεί με ένα λίγο πιο ουδέτερο και λίγο πιο κατανοητό τρόπο. Και αυτό λοιπόν το θεωρώ πολύ θετικό. Επίσης όσον αφορά τα συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα και όσον αφορά και την τελική έκθεση χαίρομαι ιδιαίτερα για την αναφορά που κάνει ο εισηγητής στη σημασία της εκπαίδευσης έτσι ώστε να βελτιωθούν οι ικανότητες, οι δεξιότητες ε, όλων σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω και δύο λόγια όσον αφορά τις δύο μελέτες τις οποίες ε, έχουμε ζητήσει. Το ένα είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία, ψήφος. Η συμμετοχή δηλαδή των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες, κάτι το οποίο είναι ένα πραγματικό φαινόμενο διαβάζω εδώ στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές τη συμμετοχή στο Βέλγιο σε σχέση με τη συμμετοχή στη Σλοβακία. Στο Βέλγιο 90% είναι το επίπεδο συμμετοχής. Ενώ στη Σλοβακία γύρω στα 30%. Βεβαίως, είναι υποχρεωτική η ψήφος ε, στο Βέλγιο. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να συγκρίνουμε την Κύπρο με το Βέλγιο. Η Κύπρο στην οποία επίσης είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στις ψηφοφορίες, παρόλα αυτά υπάρχει μία θεαματική πτώση των ποσοστών συμμετοχής. Μπορεί λοιπόν κανείς εδώ να αμφισβητήσει κάποια από τα στοιχεία αυτά είναι όμως πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη και τα αποτελέσματά της και βλέπουμε ότι είναι πολύ καθοριστικό όταν εξετάζει κανείς τα εκλογικά συστήματα. Μία μόνο χώρα, μέρος, ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εστονία, που είναι ένα εντυπωσιακό πρότυπο. Από την άλλη έχουμε την Ελβετία και την Ορβηγία, μη μέλη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, όσον αφορά την ηλεκτρονική συμμετοχή ή e participation, το θέμα των λεγόμενων πλατφόρμων ενημέρωσης συμμετοχής παρουσιάζεται πολύ συγκεκριμένα αυτό το εγχείρημα. Είναι ένας νέος καινοτόμος τρόπος συμμετοχής και βεβαίως αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον των πολιτών για τα ευρωπαϊκά θέματα, για την πολιτική σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Πρέπει να δούμε λοιπόν με πολύ ρεαλιστικό τρόπο το θέμα αυτό και βλέπουμε αυτές τις θεαματικές εξελίξεις οι οποίες θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, εισηγητή και είμαι σίγουρος ότι η έκθεση που μας ε, ετοιμάζει θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την εξαιρετική δουλειά που έκανε πάνω στο θέμα της ε, ηλεκτρονικής δημοκρατίας και θα ήθελα να ε, τον ευχαριστήσω που υιοθέτησε πολλές από τις παρατηρήσεις που κάναμε την προηγούμενη φορά. Το αρχικό κομμάτι που έχει να κάνει με την απογοήτευση των πολιτών, ε, λυπάμαι που αφαιρέθηκε. Δεν νομίζω ότι είναι ιδεολογική αυτή η δήλωση όπως υπόθηκε την προηγούμενη φορά. Νομίζω ότι αποτελεί μια σωστή απεικόνηση της κατάστασης. Εγώ μάλλον βλέπω τα πράγματα διαφορετικά από τον κύριο Πρέντα. Και να πω επίσης ότι λυπάμαι που το έγγραφο εργασίας που έχουμε μπροστά μας δεν είναι η επικαιροποιημένη εκδοχή του κειμένου. Είναι του Απριλίου. Είναι κρίμα λοιπόν που μιλάμε τώρα με βάση ένα παλαιό έγγραφο. Πάντως ε, όσον αφορά την ε, εισαγωγή πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς. Ε, πολύ σύντομα θα έχουμε το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και εδώ και μέρες ε, φαίνεται σαν να πρόκειται να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε αυτό στο κείμενο, διότι είναι μία ε, ακραία ένδειξη ότι ο, οι πολίτες νιώθουν πολύ μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν ε, ο εισηγητής ε, να συμπεριλάβει αυτό που είχε αρχικά στο κείμενο, ώστε να φαίνεται η απόψένωση και η απογοήτευση στο κείμενο. Αναφέρομαι στην εισαγωγή που τώρα πια έχει αφαιρεθεί από το κείμενο. Ο συγκεκριμένο συλλογισμό όμως πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στο έγγραφο. Στο έγγραφο λοιπόν του Απριλίου μιλάμε για αποξένωση και απογοήτευση των πολιτών. Αμφισβητούν τους εκπροσώπους τους και έχουν μειωμένη συμμετοχή στη δημοκρατία. και αποτελεί αυτό απόρριψη όχι των ε, θεσμών αλλά του ευρωπαϊκού εγχειρήματο συνολικά και δεν μιλάμε απλά για απογοήτευση, πρόκειται για οργή. Ας μην εθελοτυφλούμε. Το εγχείρημα αυτό έχει κοινωνικο-οικονομική και πολιτική ιστορία και χθες ακούσαμε πάλι για το Brexit. Ε, παλαιότερα μιλούσαμε για την έξοδο της Ελλάδας. Ε, τα δύο αυτά θέματα συνδέονται στενά μεταξύ τους. Στο κίνημα του Brexit ε, τίθενται θέματα δημοκρατίας, τα οποία δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε. Συζητιέται η κυριαρχία των διαφόρων χωρών και αυτά που υπόθηκαν, αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα συζητώνται και από αυτούς που είναι υπέρ της αποχώρησης ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει απόσταση ανάμεσα στον Δήμο και το κράτος και εκεί οφείλεται η αποξένωση και απογοήτευση των πολιτών. Βλέπουμε λοιπόν αδιαφορία των πολιτών. Είχαμε πρόσφατα μία δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία λέει ότι μετά από τρία χρόνια Πρωτοβουλία των πολιτών είναι ακόμα πολύ νωρίς να αναθεωρήσουμε τον σχετικό κανονισμό. Βλέπουμε λοιπόν από την πρόταση αυτή ότι η Κομισιόν δεν ακούει αυτό που θέλουν οι πολίτες. Δηλαδή, εργαλεία άμεσης δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι είναι πολύ νωρίς να ακούσουμε τι θέλουν να μας πούν οι πολίτες. Και εάν αναλύσουμε περαιτέρω το κείμενο, τίθεται και το θέμα του τι πρέπει να κάνουμε. Και θα ήθελα εδώ να επισημάνω το εξής. Λέμε ότι η ψηφιακή δημοκρατία θα πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση του τρόπου διακυβέρνησης και της ε, διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Αυτό θέλω να πω στον εισηγητή. Όταν μιλάμε για την κρίση, για το έλλειμμα δημοκρατίας που διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο στόχος ε, θα πρέπει να είναι όχι μόνο η διαδικασία διακυβέρνησης, ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή των πολιτών. Το θέμα δηλαδή δεν είναι πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι τα πράγματα. Το θέμα είναι πώς έχει η κατάσταση στην πραγματικότητα. Δεν θα πρέπει οι πολίτες να νιώθουν ότι τους ε, αγνοούν τα θεσμικά όργανα. Νομίζω ότι στις 10 Απριλίου είχαμε τελευταία φορά τη συζήτηση αυτή και επιμένω ότι η ψηφιακή δημοκρατία θα πρέπει να αποτελεί μια συνεχόμενη διαδικασία και όχι να ολοκληρωθεί με μία ψηφοφορία. Και η τελική μου παρατήρηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αλλάξει. Στην πρόταση αυτή έχουμε την ευκαιρία να πούμε ότι πρέπει να επιλέξουμε τη σωστή διαδικασία να έχουμε μια διαδικασία όχι από πάνω αλλά από τη βάση. Διότι αλλιώς με τη συζήτηση που έγινε για την Ελλάδα, με την συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τον Brexit, θα είναι το τέλος του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Ευχαριστώ πολύ από τους Πρασίνους. Ο κύριος Σόφλιν θα πάρει το λόγο, παρακαλώ. ο κύριος Σέφλιν μπορεί να πάρει το λόγο πριν από μένα. Ε, ε, ο κύριος Σέφλιν θα πάρει το λόγο πρώτος, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να εκφράσω κάποιους συλλογισμούς ε, σε σχέση με αυτά που μόλις είπε η κυρία Σπινέλη, τα οποία δεν συνδέονται και πάρα πολύ στενά με το έγγραφο του κυρίου ε, Χαουρέγγι, διότι πάντα θα υπάρχει απόσταση ανάμεσα στο Δήμο και το κράτος. Το πρόβλημα είναι το εύρος του χάσματος και ειδικά όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ξέρω ότι δεν είναι μέρος της ε, σημερινής συζήτησης, αλλά ήμουν εισηγητής και έχω αρκετά ε, αξιόπιστες πληροφορίες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να παγώσει το μέσο αυτό. Μπορώ να μαντέψω μόνο ποιες είναι οι αιτίες για αυτό, πάντως αυτή είναι η κατάσταση. Ε, γι' αυτό όταν ε, έρθει ο, ο ε, Αντιπρόεδρος Τίμερμανς θα αποτελέσει προτεραιότητα για μένα η, μια σχετική ερώτηση. Όσον αφορά την έκθεση που έχουμε μπροστά μας, το έγγραφο εργασίας, τέσσερις παρατηρήσεις. Εγώ θα τόνιζα πολύ περισσότερο το θέμα της ε, κυβερνοασφάλειας. Υπάρχει στο κείμενο, αλλά εγώ θα το τόνιζα περισσότερο. Δεν είμαι εμπειρογνώμονας, αλλά πόσο καταλαβαίνω εγώ το κείμενο, κάθε επίπεδο ασφάλειας μπορεί να παραβιαστεί. Αυτό είναι γεγονός στο διαδίκτυο και το έχουμε συμπεριλάβει στο κείμενο. Δεύτερη παρατήρηση. Στον ηλεκτρονικό κόσμο βλέπουμε ραγδαίες αλλαγές. Όλοι έχουμε smartphone τώρα πια, ενώ πριν τρία χρόνια δεν ήταν έτσι. Και νομίζω ότι θα θυμάστε τις γραφομηχανές. Ε, πολλοί νέοι άνθρωποι δεν έχουν δει ποτέ τους ε, γραφομηχανή. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον τρόπο που θα ξεπεραστούν οι σημερινές τεχνολογίες. Δεν έχουμε μια γραμμική διαδικασία. Αλλά η δημοκρατία, η πολιτική ζωή απαιτεί κάποιο βαθμό σταθερότητας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί κάποια αναφορά στην σταθερότητα. Θα πρέπει να παρακολουθούμε την τεχνολογία, διότι αλλιώς θα καταλήξουμε οι πολίτες να χρησιμοποιούν ε, τεχνολογίες που ε, έχουν πια ξεπεραστεί. Όσον αφορά την αναβάθμιση των ε, δεξιοτήτων, αυτό συνδέεται με τις τεχνολογικές αλλαγές που μόλις ανέφερα. Βλέπουμε μια σημαντική αλλαγή στις ε, κοινωνίες μας, ε, ενώ την Ευρώπη, τη Δύση γενικά. Βλέπουμε όχι μόνο τη γύρανση του πληθυσμού, αλλά οι σημερινοί τριαντάριδες είναι πολύ πιθανό να ζήσουν 100 χρόνια. Δηλαδή, η δημογραφική ισορροπία θα αλλάξει. Ε, θα, το, 50, ε, το 60% της κοινωνίας ε, θα είναι άνω της ηλικίας των 60 ετών. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι δυνατότητες τους, αλλά ο ρόλος του πολίτη θα απαιτεί κάποιο βαθμό τεχνολογικών δυνατοτήτων, κάτι που δεν ίσχυε στο παρελθόν. Βλέπουμε τη δουλειά που έχετε κάνει. Αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας, ε, μιας συνεχούς διαδικασίας. Ε, δεν θα υπάρξει τέλος στη διαδικασία αυτή, όπως άλλωστε δεν υπάρχει τέλος στην εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπιέ. Είναι η πρώτη φορά που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, <clears throat> παρόλο που είναι η πρώτη μου συμμετοχή σαν αναπληρωματικό μέλος αυτής της Επιτροπής. Διάβασα πριν από λίγο την έκθεση του συναδέλφου και λίγες είναι οι παρατηρήσεις που έχω να κάνω επιπλέον από αυτές που ακούστηκαν ήδη. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι, επειδή εκλέγομαι σε μια περιοχή που αντιστοιχεί στο 16% της γαλλικής επικράτειας με 9 εκατομμύρια κατοίκους, με μικρές πόλεις, με χωριά, με χωριουδάκια, όπου δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναρωτηθούμε για θέματα όπως την ε, ψηφιακή πρόσβαση και την ψηφιακή ηλεκτρονική συμμετοχή και δημοκρατία. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε καν σύνδεση στο ίντερνετ. Η δεύτερη πρόταση που κάνετε στη σελίδα 5, εκεί που αναφέρεται την πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία και το ξεπέρασμα του χάσματος. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να αλλάξουμε τη διατύπωση και να μιλήσουμε για την πρόσβαση σε περιοχές, σε εδάφη που δεν είναι πύκνο κατοικημένα και που δεν έχουν απολύτως καμία πρόσβαση. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε καν την πολυτέλεια να αναρωτηθούμε σε πολλές από τις περιοχές της εκλογικής μου περιφέρειας για το αν ή όχι θα έχουμε πρόσβαση σε αυτή την ε, ηλεκτρονική συμμετοχή. Και αν κοιτάξει κανείς ένα χάρτη θα διαπιστώσει ότι αυτοί που ψηφίζουν ακραίες πολιτικές δυνάμεις πολλές φορές είναι αυτοί που ζουν σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές ή αποκλεισμένες περιοχές. Πολλές φορές δηλαδή οι ψηφοφόροι αυτοί δεν έχουν σχέση καν με φαινόμενα σαν τη μετανάστευση. Απλώς νιώθουν απομακρυσμένοι. Πρόκειται για πολίτες που ζουν απομονωμένοι και οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση και θα ήθελαν πάρα πολύ να μπορέσουν να συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και να γίνουν ενδεχομένως και ψηφιακοί πολίτες. Ευχαριστώ πολύ κύριο Άντερσον. Ευχαριστώ. Κάτι που πιστεύω ότι θα πρέπει με πιο συγκεκριμένο τρόπο να αναφερθεί, θα βρούμε έναν τρόπο να το διατυπώσουμε εξάλλου, είναι οι ευκαιρίες, οι δυνατότητες, αυτή η ψηφιακή δημοκρατία να βοηθήσει τους πολίτες να εκφραστούν όσον αφορά την πολιτική διαδικασία και τα τεκτενόμενα. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να εκφραστούμε, αλλά το δημόσιο συμφέρον δεν είναι τόσο ισχυρό σε σχέση με τα ιδιωτικά συμφέροντα. Αν έχει κάποιος δηλαδή κάποια ειδικά συμφέροντα, αν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ομάδες πίεσης, τα λόμπι και να δαπανίσει κεφάλαια, μπορεί να αποκτήσει ένα πλεονέκτημα. Όταν όμως υπάρξει πληροφορία, επικοινωνία, η οποία θα είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη σε όλους, αυτό το σύστημα θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο παιχνίδι, πιο ίσες συνθήκες για όλους. Και αυτό θα ήταν κάτι το πάρα πάρα πολύ θετικό, πιστεύω. Τώρα, όσον αφορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία, αυτό Πιστεύω ότι παρουσιάζεται με ισορροπημένο τρόπο. Εγώ αν έγραφα αυτό το κείμενο θα έλεγα ότι πρόκειται για μια τρομερή ιδέα, αρνητικά τρομερή ιδέα. Ξέρω όμως ότι δεν συμφωνούμε όλοι όσον αφορά το θέμα αυτό. Ξέρω ότι στην Επιτροπή μας υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την ηλεκτρική ψηφοφορία και πιστεύω ότι αυτό το κείμενο παρουσιάζει με κάπως ισορροπημένο τρόπο αυτό το θέμα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσω είναι το θέμα της απάτης. Εάν υπάρχουν καταχρήσεις και εάν τελικά επικρατήσει η ιδέα ότι πρέπει να ψηφίζουμε με ηλεκτρονικό τρόπο, θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη γιατί ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους πολίτες να καταλάβουν γιατί και πώς ένα ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας είναι ασφαλές. Δεν είναι εύκολο να εξηγήσει κανείς το τεχνικό κομμάτι στους πολίτες. Και καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν ε, ερωτηματικά και ανησυχίες, αυτό θα οδηγήσει σε ακόμα ε, λιγότερη εμπιστοσύνη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να εξετάσουμε και αυτό το θέμα της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας αυτού του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας. Σε γενικές γραμμές ε, πιστεύω ότι το κείμενο είναι καλό. Τα σχόλια είναι σε πιο δευτερεύοντα συστήματα. Εδώ αναφερόμαστε παραδείγματος χάρη στις διάφορες μεταρρυθμίσεις του εκλογικού συστήματος. Αυτό όμως τι ακριβώς σημαίνει. Διαφορετικά ανώτατα όρια, κατώτατα όρια, ότι θα πρέπει να εξαλειφθούν οι πιο μικρές εκλογικές περιφέρειες, δεχομένως το σύστημα της Σουηδίας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία το οποίο εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες με περίεργο τρόπο. Για μένα αυτό δεν θα ήταν κάτι το πολύ θετικό. Θα προτιμούσα να επικεντρωθούμε στα κεντρικά σημεία αυτής της έκθεσης που είναι η ψηφιακή δημοκρατία. Και να αποφύγουμε ιδέες και προτάσεις οι οποίες μπορεί να φαίνονται πολύ ενδιαφέρουσες αλλά θα μπορούσαν να παρερμηνευθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κυρία Μπρέσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ραμόν Χάουρεγγι για αυτό το δεύτερο έγγραφο εργασίας το οποίο προφανώς δεν είναι ακόμα το τελικό κείμενο και επί του οποίου θα μπορέσουμε και εμείς καλύτερα να προβληματιστούμε. Πάντως πιστεύω ότι σίγουρα μας δίνει όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειαζόμαστε για να προβληματιστούμε. Και αντικειμενικά είναι πάρα πολλά αυτά. Και τόσο που δυσκολεύουν και την ίδια μας τη συζήτηση. Έχει όμως σημασία και είναι καλό το γεγονός ότι βλέπουμε όλη αυτή τη διαδικασία σε πολλά στάδια και πώς μπορούμε απολύτως να χρησιμοποιήσουμε τις ψηφιακές δυνατότητες που έχουμε για τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Πολλά από τα ε, όσα είπε η κυρία Σπινέλη με βρίσκουν σύμφωνοι και άλλα πάλι όχι. Αλλά έχουν να κάνουν ακριβώς με τη δημοκρατία γενικότερα, όχι μόνο την ψηφιακή. Τώρα ενδεχομένω μπορεί να βοηθούν τα εργαλεία τα ψηφιακά, αλλά λύση δεν είναι στα ευρύτερα προβλήματα της δημοκρατίας. Το το μέσον δεν είναι το μήνυμα της δημοκρατίας. Είναι ένα στοιχείο μόνο. Θα έχουμε πάντως ε, την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε μετά το Βρετανικό Δημοψήφισμα όταν θα συζητάμε και για άλλα μέσα της δημοκρατίας εκτός από το δημοψήφισμα και τα ψηφιακά. Πάντα όλα αυτά έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα ε, στα οποία έχει οριμάσει η εκτίμησή μας και η αξιολόγηση. Ο Ραμόν ονομάζει κάτι e-governance, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή μπαίνει και αυτό το θέμα του ψηφιακού χάσματος που ανέφερε ο κύριος Λαβρίο, γιατί άμα δεν λυθεί αυτό, τι να το κάνουμε, δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά έχει σημασία να έχουμε ως στόχο την καθολική ε, χρήση από πλευράς δημόσιας διοίκησης αυτών των ψηφιακών εργαλείων για να διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών. Παράδειγμα. Αν θέλει ένα ε, δημόσιο έγγραφο μπορούν να στο στείλουν επιγραμμικά ή πρέπει να στείλουν όλο το φάκελο για να είναι εντάξει η γραφειοκρατία, η δημόσια διοίκηση ότι έχει όλα τα χαρτιά ή το αντίστροφο. Θα πρέπει να είναι πιο εύκολη λοιπόν η πρόσβαση και η σχέση του πολίτη με το δημόσιο που είναι τόσο βαριά που δεν βλάπτει και λίγη απλούστευση. Πάντο, μα και που... Αναπτύσσεται λοιπόν αυτό το θέμα, εξελίσσεται ε, και ε, υπάρχει ένα τμήμα του πληθυσμού όμως που ε, αποκλείεται από αυτή την προσπάθεια, είτε για λόγους τεχνικούς, ότι δεν έχουν καλή ε, σύνδεση και το που πάνε να κάνουν μια δύσκολη ε, δουλειά ε, πέφτει, κρασάρει το διαδίκτυο και το χαλάει. Θα μπορούσαν όμως όλοι να υποφελούνται από αυτή τη δυνατότητα αν ήταν καλή η κάλυψη. Λοιπόν, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι κάτι το σημαντικό και το σωστό. Ας πούμε ότι ξεπερνάμε το ψηφιακό χάσμα, το τεχνικό και το πολιτισμικό και της νοοτροπίας. Εκεί ανοίγει μια λεωφόρος για χρήση για πιο περίπλοκες ακόμα και πιο δύσκολες ε, ε, διαδικασίες ε, και διεργασίες της δημοκρατικής ζωής. Ο Ραμόν Χαοριγκή το χαρακτηρίζει όλο αυτό ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Το είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι 28 χώρες, ελπίζω και αύριο να είμαστε 28 και να μην πάθουμε καμία ζημιά, ε, με τόσα εκατομμύρια ε, κατοίκων να μπορούν να λένε τη γνώμη τους, να γίνεται δημόσια διαβούλευση από τον απλό πολίτη μέχρι τους stakeholders, τους ενδιαφερομένους και ενεχομένους. Για να γίνει αυτό μόνο ε, online γίνεται. Ακόμα είμαστε σε πολύ πειραματικό στάδιο. Πάντως υπάρχει έδαφος να αναπτυχθεί η δυνατότητα διαβούλευσης δημόσιας, ακόμα και η δυνατότητα κατανόησης ε, των διαφόρων ε, καταστάσεων και προτάσεων. Γιατί θα πρέπει ο πολίτη να κάνει τη φωνή του να ακούγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην επιβάλλονται διάφορες αποφάσεις σε του. Καλύτερη χρήση λοιπόν χρειάζεται αυτών των εργαλείων και ε, για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για να είναι πιο εύκολη η διαδικασία και πιο εύχρηστη. Όλα αυτά εντάσσονται στο συγκεκριμένο θέμα. Ένα τελευταίο που θέλω να πω για την ηλεκτρονική ψηφιακή δημοκρατία. Αυτό τώρα είναι πιο περίπλοκο. Για ποιο λόγο. τα ψηφιακά εργαλεία, πώς να το πω, τουλάχιστον υποθετικά, επιτρέπουν κάποιους τρόπους άμεσης δημοκρατίας που κατά κάποιο τρόπο συγκρούονται με τις κλασικές αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Έχουμε μια μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη, δεν ξέρω στον κόσμο, αλλά νομίζω και στον κόσμο είναι μοναδικό, αντιπροσωπευτικής και άμεσης δημοκρατίας ε, που λειτουργεί πάνω κάτω καλά. Αυτό είναι η Ελβετία. Στην Ελβετία υπάρχουν κανονικοί δημοκρατικοί θεσμοί αντιπροσωπευτικοί και ισχυροί, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα σύστημα άμεσης δημοκρατίας, περίπλοκο, πολύ καλά οργανωμένο, που επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν ε, και αυτό κάπως παντρεύεται μετά με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και εκφράζει τη γνώμη του λαού. Δηλαδή μέχρι σημείο που μπορεί να αλλάξει το σύστημα με νομοθετική πρωτοβουλία, που αυτό είναι και μεγάλη υπόθεση. Πάντως λειτουργεί αυτό. Είναι μια χώρα που έχει βαθιά ριζωμένη την δημοκρατική παράδοση, αλλά και ακόμα και εκεί ε, υπάρχει δυνατότητα ε, ενδεχόμενο εκτροπής, γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Ε, ο λαϊκισμός αυξάνεται. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό των περιόδων κρίσεων. Μετά από κάθε οικονομική κρίση ε, οργιάζει ο λαϊκισμός και υπάρχει φόβος για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία κινδυνεύει όταν έχουμε μεγάλες οικονομικές κρίσεις, όπως αυτή που ζούμε και δεν έχει ακόμα τελειώσει, δεν έχουμε γλιτώσει. Ακόμα λοιπόν και στην περίπτωση της Ελβετίας που είναι τόσο καλά ε, στημένο το σύστημα, δηλαδή λειτουργεί, ε, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα και πολύ επικίνδυνες συνέπειες όταν τα πράγματα σφίγγουν. Όταν πάνε όλα καλά, ο λαός αποφαίνεται. Με τρόπο φρόνιμο και λογικό. Ε, όταν σκουραίνουν, μπορεί να εκφραστεί ο λαός ε, και με τρόπο που να ε, απειλεί και το habeas κόρπους και τα ατομικά δικαιώματα. Αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να το σκεφτούμε όταν αναπτύσσουμε εργαλεία ηλεκτρονικής δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε μια ήπειρο που έχει διαφορετικές παραδόσεις. Αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίσει όμως ε, από το να πειραματιστούμε, να το προσπαθήσουμε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Η κυρία Σπινέλη προηγουμένως μίλησε ε, για την τοπική αυτοδιοίκηση, για το bottom-up το bottom συγγνώμη, που είναι από, από κάτω προς τα πάνω η προσέγγιση από τη βάση στην κορυφή και εγώ από την τοπική αυτοδιοίκηση προέρχομαι. Αλλά δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε έρχεται από το λαό ε, είναι εντάξει αν γίνεται μόνο online χωρίς τα διάφορα φίλτρα για να διηθούν τη συζήτηση, την άμεση συζήτηση και την άμεση διαβούλευση. Να ακούγονται και οι μειονότητες και οι απόψεις της μειοψηφίας, αλλά προσοχή. Αυτό μπορεί να έχει και πάρα πολύ επικίνδυνα και στρεβλά αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτή η ηλεκτρονική δημοκρατία μπορεί να ξεφύγει καμιά φορά. Αλλά τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα πρέπει να τα έχουν αυτά υπόψη του όσο και αν είναι προβληματικά. Θα πρέπει να εργαστούμε προ την κατεύθυνση αυτή και θα ήταν και ενδιαφέρον να γίνει μια προσπάθεια και να προωθηθεί. Θα πρότεινα στο Ραμόν, στο έγγραφο που προετοιμάζει, ενδεχομένως να σκεφτούμε, να κοιτάξουμε να δούμε με ποιο τρόπο οι μηχανισμοί άμεσης δημοκρατίας μπορούν να λειτουργήσουν με νέα εργαλεία που δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί και δεν έχουμε τον πλήρη έλεγχό τους. Και τα προβλήματα δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα. Προσοχή λοιπόν. Η κοινωνιολογία της συμπεριφοράς των μαζών μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα. Ε, και η δεκαετία του 30 ξέρουμε πολύ καλά τι δείχνει και τι σημαίνει για ε, μαζικά ανεξέλεγκτα κινήματα. Και αυτά μπορούν να γεννηθούν και online ακόμα και ακόμα πιο γρήγορα και με λιγότερα φίλτρα, λιγότερες δυνατότητες ελέγχου και επαλήθευσης. Αυτά με απασχολούν Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν μπορεί κανείς να εμποδίσει τα εργαλεία αυτά να αναπτύσσονται. Ας το δοκιμάσουμε για να δούμε πώς λειτουργούν και πώς μπορούμε να εγγυηθούμε βασικά στοιχεία της δημοκρατίας. Που είναι η αντιπαράθεση των απόψεων, δεν μπορεί κανείς να αποφασίζει χωρίς να ρωτήσει και να διαβουλευτεί, αλλά ταυτόχρονα να γίνονται σεβαστές και οι που είναι άλλη βασική και θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας. και δεν είναι πάντα δεδομένο αυτό. Αυτό είναι ο βασικός κίνδυνος. Και αρχίζει να αναδύεται και να διαφαίνεται. Είναι πολύ σημαντικό όμως να προβληματιστεί το Κοινοβούλιο, γιατί όχι. Ελπίζω να γίνει αυτή η συζήτηση. Η δική μας Επιτροπή είναι ο εμπνευστή, η κινητήρια δύναμη. Δεν είναι τελευταία φορά που θα τα συζητήσουμε αυτά αλλά είναι σημαντικό να γίνει αυτή η προσπάθεια, κάποιος να κάνει την αρχή. Ας το δοκιμάσουμε και να δούμε, να το προτείνουμε πώς θα προχωρήσει για να καταλάβουμε και όλα τα προβλήματα που μπορεί να είναι και τεχνικά και πολιτικά κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εισηγητή καθώς και τους σκιώδης εισηγητές. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στην εξέβριση συνένεσης. Προφανώς θα πρέπει να εξετάσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα έχουν στόχο την ευρύτερη πολιτική συμμετοχή. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, Συγγνώμη, ξέχασα να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα μόνο να πω το εξή πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους. Ήταν πάρα πολύ εύστοχα όλα αυτά που είπαν. Πολύ πλούσια συζήτηση, πολύ έντονη, με πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις. Τις σημειώνω όλες και του κυρίου Σόφλεν και του κυρίου Πρέντα και του άλλου συναδέλφου του κυρίου Λαβριέ από το ΕΛΚ. Και ε, προφανώς αυτά ε, θα βελτιώσουν ε, κάποιες από τις ιδέες μου, θα τα συμπεριλάβω στη σκέψη μου. Επ' ευκαιρία, σήμερα πήραμε δύο έγγραφα από την Υπηρεσία Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά, παρακαλώ να τα κοιτάξουμε. Και επίσης θα συμπεριλάβω ιδέες από αυτά στο πρώτο σχέδιο έκθεσης που θα έρθει το Σεπτέμβριο και θα είναι εμπλουτισμένο με τις ιδέες που προτείνατε και που λέει και το έγγραφο εδώ. Δεν μπορώ να κάνω συζήτηση ουσίας με την Μπάρμπαρα Σπινέλη γιατί δυστυχώς δεν έχουμε εδώ το χρόνο. Δηλαδή και το χώρο, το νέο κείμενο που φέραμε σήμερα είχε περιορισμούς. Μπορεί να λύνει κάποια θέματα από τα όσα ίδια αναφέρει. Είπε η κυρία Σπινέλη ότι η έκθεση αυτή θα μπορούσε να ασχοληθεί με τις βαθιές ρίζες της απαξίωσης της πολιτικής των αντιευρωπαϊκών αισθημάτων των πολιτών κτλ. Εγώ με πολύ μεγάλη χαρά θα τα συζητούσα αυτά τα πράγματα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αλλά θα σας παρακαλούσα και θέλω να το πω ιδιαίτερα στην Μπάρμπαρα να ακούσετε ότι η έκθεση αυτή έχει λιγότερη φιλοδοξία δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε όλα τα προβλήματα της δημοκρατίας με την τεχνολογία. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και συνετοί, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, είπε και η Μερσέντες Μπρέσο. Πιθανότατα, όχι καθόλου πιθανότατα, είμαι βέβαιος ότι συμφωνούμε Μπάρμπαρα, αλλά τα προβλήματα του αντιευρωπαϊσμού, ε, του νέου εθνικισμών στην Ευρώπη, όλα αυτά που αναδύονται ε, στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η διαμαρτυρία εντό εισαγωγικών ε, όχι στην Ευρώπη, Brexit, η αντίδραση αυτή των πολιτών, όλα αυτά είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ θα ήθελα ταπεινά να πω ότι η έκθεσή μου έχει ως στόχο απλώ να βελτιώσει τη δημοκρατία μας ως προς το ηλεκτρονικό σκέλος με τις τεχνολογίες, τις ψηφιακές αυτές και της επικοινωνίας. Δυστυχώς, την άλλη εβδομάδα, ανάλογα με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αυτές οι συζητήσεις θα μας κατακυριεύσουν και θα μας ξεπεράσουν, αλλά θα τις κάνουμε άλλη ώρα, όχι αυτή τη στιγμή. Θα συμπεριλάβω και τις δικές σου ιδέες, Μπάρμπαρα, στην αιτιολογική έκθεση ε, της έκθεσης μου, όχι στο, στα άρθρα ας πούμε, αλλά στην αιτιολογική έκθεση μπορώ να τα αναφέρω αυτά. για είναι πιο πολιτική η τοποθέτηση. Τελειώνω, Πρόεδρε. Επί της ουσίας τι θέλουμε. Να βρούμε μια ισορροπία, πολύ ωραία το είπε κύριος Άντερσον, ανάμεσα στις ευκαιρίες και τους κινδύνους, τα ρίσκα. Γιατί η συζήτηση αυτή, πώς γίνεται, ανάλογα με το που μπαίνει το κέντρο βάρους, ε, παίρνει άλλη στροφή η έκθεση. Αν το παρακάνουμε με, τα, ε, με τους κινδύνους, υποτιμούμε τις ευκαιρίες. Από την άλλη, αν τα παρουσιάσουμε όλα ρόδινα, τι ωραίος κόσμος, χωρίς να αξιολογήσουμε και τους κινδύνους που έχει το χάσμα αυτό το ψηφιακό και το εδαφικό και όλα αυτά, η χρήση ε, που έχει κινδύνους, δηλαδή, το πώς θα κάνουν κατάχρηση των πληροφοριών ορισμένη. Εάν δεν βρούμε αυτή τη χρυσή τομή, η έκθεση κινδυνεύει να είναι όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος. Εγώ θέλω να προκαλέσω και μια συζήτηση. Το είπε και ο κύριος Σόφλη, που μόλις αρχίζει τώρα και θα συνεχιστεί πιθανότατα. Μίλησε για την τεχνολογική εξέλιξη και θυμάμαι ότι διάβαζα πριν από λίγο καιρό μια έκθεση που έλεγε ότι τώρα γεννιούνται παιδιά που θα ζήσουν 140 χρόνια. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι δεν ξέρουμε ακόμα πολύ καλά πού το πάει η τεχνολογία και τι κόσμος μας περιμένει με την τεχνολογική αυτή επανάσταση που εξελίσσεται με γεωμετρική πρόοδο. Συγγνώμη Πρόεδρε, απλώς ήθελα να πω ότι όλες οι ιδέες που ακούσαμε θα τις συμπελάβουμε για να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα έγγραφο το οποίο ελπίζω όλοι να υποστηρίξουν. Τροπολογίες θα μπορέσετε φυσικά να κάνετε και πολύ συγκεκριμένες όλα τα μέλη και όλες οι πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πιστεύω ότι ο αντίκτυπος της έκθεσης αυτής θα είναι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Το χρονοδιάγραμμα 29 Σεπτεμβρίου, εξέταση του σχεδίου έκθεσης. 13 Οκτωβρίου, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Προχωρούμε τώρα στο σημείο 9. Δημοσιονομική ικανότητα για την Ευρωζώνη. Έχουμε να συζητήσουμε την... το σχέδιο της γνωμοδότησης καθώς και τις τροπολογίες. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο. Ο κύριος Παύλο Ραγγέλ θα αντικατασταθεί από τον κύριο Πρέντα. Του δίνω λοιπόν το λόγο. So, um, I... Ευχαριστώ πολύ. Θα, θα σας διαβάσω το κείμενο που έλαβα από τον συνάδελφό μου, τον κύριο Ραντζέλ. Έχουμε λοιπόν σχέδιο γνωμοδότηση τη ΑΦΚΟ που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Προπολογισμών ε, τον Απρίλιο για ανταλλαγή απόψεων. Τονίζει ότι η δημιουργία δημοσιονομικής ικανότητας για την Ευρωζώνη είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η ΟΝΕ. Και ως προς το περιεχόμενο λέει ότι στο σχέδιο έκθεσης εκφράζει την υποστήριξη για ανάπτυξη δημοσιονομικής ικανότητας στην Ευρωζώνη ε, και αναφέρεται στο άρθρο 310, 311 και 312 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις δυνατότητες ε, που προβλέπονται σε αυτά τα άρθρα, αλλά και σε άλλα άρθρα όπως είναι ε, αυτά του κανονισμού για, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχουν ε, κάποια πρωτόκολλα που προβλέπουν επίσης ε, και τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ήταν 7 Ιουνίου και έχουν υποβληθεί 86 τροπολογίες και έχουν σταλεί για μετάφραση. Το συμπέρασμα του κυρίου Ραντζέλ έχει ω εξή. Λέει ότι θα ήθελε να ευχαριστήσει όλου του συναδέλφου που έχουν υποβάλει τροπολογίε για τη δουλειά που έχουν κάνει και υπόσχομαι ότι θα τι εξετάσω όλε και θα προσπαθήσω να καταλήξω σε συμβαστικό κείμενο που να πληρεί τις προσδοκίες ε, των περισσότερων. Ε, στις 12 ε, Ιουλίου προβλέπεται η ψηφοφορία στην ΑΦΚΟ, γι' αυτό θα σας στείλω κείμενο όσο γίνεται πιο γρήγορα, σεβόμενο στις προθεσμίες. Ευχαριστώ. Έχουμε την κυρία Μπέρες για την Οικονομική Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σε όλα τα μέλη της ε, Επιτροπής ΑΦΚΟ που υπέβαλαν τροπολογίες. <clears throat> Έριξα μια ματιά και βεβαίως ε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Φαντάζομαι ότι ο κύριος ε, Ράντζελ θα καταφέρει να παρουσιάσει με ισορροπημένο τρόπο τη θέση της Επιτροπής. Κάποιες από αυτές ε, δεν μπορεί να γίνουν ε, αντικείμενο συζήτησης, καθότι παραδείγματος χάρη αμφισβητούν την ύπαρξη του κοινού νομίσματος με την έννοια ότι δεν μπορεί να ενσωματωθούν σε καμία απολύτως συμβαστική πρόταση. Το θέμα επίσης της οργάνωσης του εσωτερικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η συνεισφορά της ε, Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Υπάρχει μία σειρά τροπολογιών και βεβαίως θα πρέπει εδώ να επιλεγούν αυτές που εκπροσωπούν την θέση της Επιτροπής ΑΦΚΟ. Όσον αφορά το άρθρο 13, και εδώ πιστεύω ότι θα μπορέσει να είναι χρήσιμη η πρόταση αυτή για τη συζήτησή μας και από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα μπορέσει να υπάρξει και συζήτηση γύρω από την έννοια του Δημόσιου Ταμείου. Αυτή η ιδέα υπάρχει στην ε, έκθεση και έχω την εντύπωση ότι από την αρχή της συζήτησης για την έκθεση αυτή με τον ε, κύριο Μπέγκε έχουμε επεξεργαστεί την ιδέα είτε ενός ε, Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου είτε ενός Ευρωπαϊκού Δημόσιου Ταμείου η επιλογή θα πρέπει να γίνει. Εμείς πάντα επιλέγουμε μάλλον την κοινοτική μέθοδο. Ίσως αυτό θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε τη μία από τις δύο αυτές ε, προτάσεις. Τελικά λοιπόν μάλλον, μάλλον βλέπω επικρατέστερη την επιλογή του Δημόσιου Ταμείου. Κάτι άλλο για το οποίο θα πρέπει να διαλέξουμε είτε θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση της συνθήκης είτε όχι. Βεβαίω εσείς είστε αρμόδιοι εδώ, πολύ περισσότερο από εμά από την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Όμως, σίγουρα θα πρέπει να επεξεργαστούμε τις δυνατότητες που έχουμε εδώ, δεν είναι μόνο η δική σας έκθεση, η, αυτή εδώ η έκθεση η οποία θα υιοθετηθεί, υπάρχουν ταυτόχρονα και άλλες εκθέσεις. Και κάτι άλλο που σίγουρα δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε είναι οι συνέπειες της συμφωνίας του Φεβρουαρίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Στα πλαίσια αυτής της ε, συζήτησης είδαμε ότι το ευρώ, μοναδικό νόμισμα, ενιαίο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτι που αποτελεί αντικείμενο της ε, συμφωνίας αυτής του Φεβρουαρίου και το λέω με διπλωματικό τρόπο. Σίγουρα και εδώ θα πρέπει να εκφραστεί η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Αλλά πιστεύω ότι με τον κύριο Ρέγκελ και τον ε, Μπέγκε θα πρέπει να συνεχίσουμε την ε, συζήτησή μας. Αυτές είναι οι πρώτες μου σκέψεις ε, έχοντας διαβάσει τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπρέσο είναι εδώ. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Είμαστε μόνο τρεις παρόντες. Η ποσότητα δεν έχει σημασία, η ποιότητα μας ενδιαφέρει, κυρία Μπρέσο. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές και έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για μια έκθεση η οποία έχει σχέση με την έκθεση του κυρίου Μπρόκ και της κυρίας Μπρέσο για την Ευρωζώνη. Η ψηφοφορία λοιπόν θα λάβει χώρα στις 12 Ιουλίου, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και στις 26 Σεπτεμβρίου στην επί αρμόδια Επιτροπή. Επιτροπή Προϋπολογισμού και Επιτροπή ΕΚΟΝ. Δύο αρμόδιες επί Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το, στο σημείο 10 Ευρώπη για τους πολίτες. Εδώ σήμερα αναφερόμαστε στην περίοδο 2014-2020 δύο μέρη 14-15 προκτήγει για τις που αφορούν το 2014 και το 2015 και το πρόγραμμα καλύπτει δύο βασικούς τομείς. Πρώτον, κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιστορικό κομμάτι, πολυμορφία και η προβολή των ε, Ευρωπαίων πολιτών καθώς και τη συμμετοχή τους ε, στην ε, Ευρώπη. Εγώ θα ήθελα εδώ να σας πω ότι έχω αναλάβει την γνωμοδότηση για την Επιτροπή Πολιτισμού και σήμερα νομίζω ότι απλώς μπορούμε να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η γνωμοδότησή μας θα πρέπει να είναι συνεκτική, σύντομη και να αφορά κυρίως πτυχές που αφορούν τις ε, δικές μας αρμοδιότητες. Το μέλλον της δημοκρατίας, συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών καθώς και η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γνωμοδότηση αυτή δεν θα πρέπει να περιέχει μόνο την ε, εφαρμογή για τα έτη 2014 και 2015 αλλά και κάποιες συστάσεις για τα σημεία αυτά που είναι αρμοδιότητας ε, της Επιτροπής μας θα γίνουν κατά κάποιο τρόπο θεματικές συστάσεις όσον αφορά την ανάπτυξη της συμμετοχής. Θεωρούμε σε κάθε περίπτωση ότι ακριβώς επειδή είχαμε τη συζήτηση για την πολιτική συμμετοχή, για την ηλεκτρονική δημοκρατία και την προσπάθειά μας να υπάρχει μεγαλύτερος αντίκτυπος ε, όσον αφορά τα θέματα της παιδείας, της επικοινωνίας, της ε, κατάρτισης. Τα θέματα λοιπόν που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής ΑΦΚΟ θα πρέπει να μας ε, απασχολήσουν περισσότερο, ιδιαίτερα για τα επόμενα χρόνια. Στις 29 ε, Σεπτεμβρίου θα συζητήσουμε για το σχέδιο γνωμοδότησης. Στις 11 Οκτωβρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι τροπολογίες και τον Νοέμβριο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή, θα λάβει χώρα ψηφοφορία στην Επιτροπή ΚΑΛΤ και στις 5 Δεκεμβρίου η τελική ψηφοφορία. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο? Δεν βλέπω κανέναν. Συμφωνήσαμε και για το χρονοδιάγραμμα και περνάμε στο σημείο 11. Η κυρία Μπρέσο. Madame Fabre, merci. thank you. S'il vous plaît, Madame Ναι. Α, πληθύναμε, λέει η κυρία Μπρέσο. Λοιπόν, ποιο μικρόφωνο να πρωτοπάρω. Αυτό. Έχουμε μετάφραση από τα ρουμανικά. Μπορώ να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, βεβαίω. Μουλτσουμέσκ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Ε, μετά το δημοψήφισμα ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να σκεφτούμε πώς αντιμετωπίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένοι πολίτες θεωρούν ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι το απόμακρο όσο και άχρηστο και αυτό εμφανίζεται τώρα όλο και περισσότερο σε διάφορα κράτη-μέλη. Ε, τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Γι' αυτό αναπτύσσονται διάφορα κινήματα αντιευρωπαϊκά. Άρα το πρόγραμμα αυτό έχει τεράστια σημασία. Το πρόγραμμα αυτό η Ευρώπη για τους πολίτες ε, γεννήθηκε το 2006 και έκτοτε χαίρομαι που έχουν χρηματοδοτηθεί ε, πολύ περισσότερα έργα. Ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις πολλέ έχουν ε, αρχίσει προσπάθειες, project και έργα. Αυτό σημαίνει ότι ε, συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες. Η αδερφοποίηση πόλεων είναι ένα πολύ καλό τρόπο ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αυτό ε, επέτρεψε να δημιουργηθούν πάγιοι δεσμοί και ισχυροί μεταξύ διαφόρων πόλεων και πολιτών ο προϋπολογισμός εκεί δεν αρκεί, μάλλον θα πρέπει να αυξηθεί για να έχει και περισσότερα αποτελέσματα, να πιάνει και περισσότερο τόπο. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει ε, κρίσιμο πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σφυριλατηθεί μια πραγματική ευρωπαϊκή ταυτότητα εάν θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες να αισθάνονται ότι τους ε, αφορά το πολιτικό αυτό εγχείρημα και όλες οι ε, ε, επιτυχίες, τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προβάλλονται, να τα γνωρίζουν οι πολίτες. Επίσης, το πρόγραμμα να είναι πιο εύκολο στη χρήση του, να έχουν πρόσβαση οι πολίτες, η κοινωνία τους, η τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, προσβλέπω στην καλή συνεργασία με τον εισηγήτη και περιμένω και το σχέδιο έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, και τώρα... Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να μιλήσει για αυτό το θέμα. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα ζητήματα. Και με κοινέ προσπάθειες θα ε, καταλήξουμε σε μια καλή γνωμοδότηση. Συμφωνώ και εγώ ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση και να αυξηθούν και οι πόροι ε, αρκεί να δει κανείς, ε, να ρίξει μια ματιά στην εφαρμογή του προγράμματος και θα καταλάβει ότι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνουν περίπου 100% των κονδυλίων που ζητούν, αλλά η συμμετοχή δεν είναι ισχυρή ε, ε, των κυβερνητικών δομών. Οι μη κυβερνητικέ δομέ αξιοποιούν αυτέ τι δυνατότητε και θέλω και η αρχή τη επικουρικότητα να ισχύει και εδώ. να ενισχύεται η διαφορετικότητα, να λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά η εκάστοτε εθνική και τοπική και περιφερειακή πραγματικότητα. Όπως σας είπα, έχουμε συζητήσει ήδη το χρονοδιάγραμμα και το επόμενο βήμα πλέον τώρα είναι η συζήτηση του σχεδίου έκθεσης στις 29 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ και προχωρούμε στο σημείο 11, το οποίο είναι και το τελευταίο για σήμερα πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασκεί το δικαίωμα εξέτασης. Τώρα έχουμε μια περίπλοκη κατάσταση Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει ακόμα αρχίσει τις εργασίες του για το θέμα αυτό. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο συνεδριάσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συγγετής είναι ο Ραμόν Χάουρεγγι. Θα τον παρακαλούσα να μας δώσει μια σύντομη εξήγηση της κατάστασης που επικρατεί και τι μας συστήνει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Διότι με έχετε ήδη ακούσει προηγουμένως για αυτό το θέμα πολλές φορές. Και επίσης θέλω να πω στην Επιτροπή τι έγινε. Σήμερα το πρωί συνεδρίασαν οι συντονιστές με την πρόεδρο μας την κυρία Χιούμπνερ για να εξετάσουμε την πρόταση που κάναμε εμείς οι Σκιώδης και εγώ ως εισηγητής για το θέμα. Θέλω να σας πω μόνο το εξής. Ενάμιση χρόνο μετά την αρχική προσπάθεια που ξεκίνησε η Επιτροπή μας, τις προσπάθειες να βρει μια συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, για να δούμε τι κανόνες διέπουν τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνει εξεταστικές επιτροπές. Ενάμιση χρόνο μετά λοιπόν δεν έχουμε καταφέρει να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις ούτε με το Συμβούλιο ούτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μεγάλο βαθμό διότι το Συμβούλιο το ερμηνεύει ως εξή. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον να το πω αλλιώς, εάν δεν διατρανώσει τη βούλησή του το Κοινοβούλιο να αλλάξουν τα άρθρα εκείνα που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και πολιτικά και νομικά από πλευρά του Συμβουλίου δεν μπαίνουν καν στη συζήτηση. Οι σκιώδεις ηγητές λοιπόν και ο υποφαινόμενος αποφασίσαμε να φέρουμε το θέμα ε, αυτό στους συντονιστές και στην πρόεδρο της ΑΦΚΟ να κάνουμε μια πρόταση για να προχωρήσουμε σε πολιτική δράση. Εγκρίναμε τέσσερα πράγματα λοιπόν και θα τα συνοψίσω πάρα πολύ γρήγορα. Τα είπαμε και το πρωί στη συνεδρία των συντονιστών. Είναι τα εξή. Πρώτον, επιστολή διαμαρτυρία στον πρόεδρο Σούλτ. Η πρόεδρο μα, η κυρία Χιούμπνερ, να την αποστείλει αυτή, που να διατρανώνει τη δυσφορία μα και, και τη διαμαρτυρία μας γιατί μπλοκάρουν το διάλογο και τις διαπραγματεύσεις και η Κομισιόν και το Συμβούλιο, ενώ οφείλουν να προχωρήσουν σε διάλογο. Είναι υποχρέωσή τους, δεν είναι στη διακριτική τους ευκαιρία. Θα πρέπει να έχουν μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα θέμα κανονισμού. Ε, λοιπόν, η κυρία Χιούμπνερ θα στείλει αυτή την επιστολή στον πρόεδρο Σούλτς, όπως είπαμε εκφράζοντας τη διαμαρτυρία μας και τα παράπονά μας και ζητώντας πολιτική απάντηση από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Δεύτερον, αποφασίσαμε να συγκληθεί συνεδρίαση της Επιτροπής μας παρουσία του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε οι ύπατοι εκπρόσωποι ε, Συμβουλίου και Επιτροπής να μας ενημερώσουν ε, σε σχέση με το αίτημά μας αυτό. Ελάτε να τα συζητήσουμε τους λέμε και στη συζήτηση αυτή μπορούν να συμμετέχουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και τέλος, μάλλον τρίτον, συμφωνήσαμε να διαβιβάσουμε στην Ολλανδική Προεδρία όπως είχαμε δεσμευτεί η κυρία Χούμπνερ και εγώ σε συνεδρίαση που είχαμε με τον πρέσβη των κάτω χωρών για αυτό το θέμα. Να διαβιβάσουμε, έλεγα, ένα κείμενο στην Ολλανδική Προεδρία, ένα non-paper, όχι επίσημο έγγραφο, όπου θα εμφανίζονται οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η διάθεσή του, προθυμία του να αλλάξει κάποια άρθρα ε, από τον κανονισμό για να ε, μπορέσει να πάρει πιο εύκολα εντολή διαπραγματευτική το Συμβούλιο. Και τέλος, ε, εάν οι νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου μας το ε, συστήσουν, δεν θα διστάσουμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο για να το υποχρεώσει να έρθει σε διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε το θέμα και που μας ε, εξηγήσατε τις τέσσερις δυσκολίες που αναφέρθηκαν και κατά τις συνεδρίες των συντονιστών. Δεν βλέπω να βρίσκεται εδώ κανένας από τους κοιόδης εισηγητές. Πρόκειται λοιπόν για μια προσπάθεια να ξεμπλοκάρει η κατάσταση. Είπατε ότι το Σεπτέμβριο μετά τις Ελληνές διακοπές θα ξανασυναντηθούμε και θα έχουμε συνάντηση της Επιτροπής μας με εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου και ελπίζουμε ότι με βάση την πρωτοβουλία μας θα μπορέσουν να προχωρήσουν πάλι τα πράγματα. Κατόπιν έχουμε τα διάφορα. Υπάρχει καμία παρατήρηση, όχι. Τότε σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι καλό απόγευμα. Λήξη της συνεδρίασης.